εγκρίθηκαν σύμφωνα με την κανονική νομοθετική διαδικασία και οι οποίες θα δημοσιευτούν. Δύο γραπτές δηλώσεις, κυρίες και κύριοι, εγκρίθηκαν από την πλειοψηφία των μελών του Κοινοβουλίου πρόκειται για το 26 του 2012 για το Global Zero για την βαθμιαία κατάργηση των πυρηνικών σε όλο τον κόσμο. Μπουτικόφε Μπαλάζα, Βαλέσσα, Κρόνμπεργκερ, Σιλβέστρη και Τσέμκε. Επίση, η παριθμόν 28 του 2012 για μια πρωτοβουλία για την δημιουργία ε, Ευρωπαϊκή ημέρα κατά τη ε, βία στα σχολεία. Κομουτσάκος, Άλβαρο, Αντζελίλη, Μπαντία, Ικουτσέτ και Τέιλορ, ε, οι συντακτέ. Οι δηλώσεις αυτές θα συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης με τις σχετικές υπογραφές. Ε, μου αναφέρεται ότι ο κύριος Βαλέσα και ο κύριος Κομουτσάκος θέλουν το λόγο. Καταρχάς ο κύριος Βαλέσα για την 26-2012 για τον Global Zero. Έχετε το λόγο κύριε συνάδελφε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Global Zero Action Plan με το Global Zero ε, Action Plan είναι μια πρωτοβουλία την, την οποία υποστηρίζουμε. Ε, Τέτοιε πρωτοβουλίε προκαλούν μεγάλη εμπιστοσύνη και είναι σημαντικό όλοι να τι υποστηρίξουμε. Όλοι να επιδιώξουμε τον σκοπό αυτό τη ενημέρωση για τα πυρηνικά όπλα. Πρόκειται για ένα σαφές μήνυμα ότι τα ατομικά και πυρηνικά όπλα αποτελούν ένα απομεινάριο του παρελθόντος και δεν έχουν καμία θέση στο σημερινό κόσμο. Αυτό θα πρέπει να μεταδώσουμε ως μήνυμα. Επιπλέον, βλέπουμε ότι τα όπλα αυτά ενδεχομένως να καταλήξουν σε λάθος χέρια. Αυτό θα ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο. Θα πρέπει λοιπόν να απαλλαγούμε από τα πρινικά όπλα και μόνο τότε θα είμαστε ασφαλείς. Προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί να συμβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση αν σταθούμε άπρακτοι, θα είμαστε συνυπεύθυνοι σε ό,τι συμβεί. Το οφείλουμε στο εκλογικό μα κοινό. Θα πρέπει να ταχθούμε υπέρ τη κατάργηση των πυρηνικών. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρο. Ευχαριστώ και τώρα το λόγο έχει για την υπαριθμόν 28 ο συνάδελφο Κουμουτσάκο. Πείτε, Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν τρει εβδομάδε, η Καρολίνα δεκατετράχονη μαθήτρια από την ιταλία έβαλε τέλος στη ζωή της. δεν άντεξε την ψυχολογική πίεση εξαιτία προσβολών και εκφοβισμού από συμμαθητές της. δεν είναι το μόνο ούτε το πρώτο από τα τραγικά θύματα ενός νοσηρού φαινομένου που τα τελευταία χρόνια αυξάνεται επικίνδυνα σε συχνότητα έκταση και ένταση. οι δραματικές κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης θρέφουν το φαινόμενο της ψυχολογικής λεκτικής και σωματικής βίας μεταξύ μαθητών. η ανωνυμία του διαδικτύου δίνει νέε διαστάσει στο φαινόμενο. Το κάνει ακόμα πιο δηλητηριώδε, ακόμα πιο επικίνδυνο. Η πρόληψη είναι ο ασφαλέστερο τρόπο αντιμετώπιση. Προποθέτει όμω ενημέρωση και γνώση. Αυτό είναι ο σκοπό τη πρόταση για την καθιέρωση Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του φαινομένου τη ενδοσχολική βία και του εκφοβισμού που υιοθετήθηκε από την πλειοψηφία των συναδέλφων. Στόχο μα ούτε ένα μαθητή θύμα ενδοσχολική βία και εκφοβισμού. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη ιδιαίτερα εκείνους που ήταν δίπλα μου από την αρχή αυτής της πρωτοβουλίας. Σήμερα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κερδίσαμε μια μάχη. Θα κερδίσουμε και τον πόλεμο. Σας ευχαριστώ κύριε Κουμουτσάκη. Κυρίες και κύριοι, σας παρακαλώ τώρα να με προσέξετε μια στιγμή σε ό,τι αφορά τις δύο αυτές δηλώσεις. Θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή στο εξής. αποφασίστηκε, μάλλον ε, σε ό,τι αφορά την Ολομέλεια, μία αλλαγή σε ό,τι αφορά τις γραπτές δηλώσεις, τις γραπτές διακηρύξεις. Από την εμπειρία, να σας πω, επειδή είμαι πολλά χρόνια το πέρα στο Κοινοβούλιο, τέτοιες αλλαγές είναι κάτι που γνωρίζουν οι συνάδελφοι ότι συνεπάγεται μια χρονική καθυστέρηση και ως εκ τούτου επειδή πάντα λαμβάνουμε επερωτήματα καταλήξαμε σε μία απόφαση το, την οποία και υπεψήφισε πλειοψηφικά το Κοινοβούλιο. Και σε αυτά συγκαταλέγεται και το ότι δεν ε, στέλνεται έδρανα πλέον από τα οποία κάνουν τις σχετικές δηλώσεις οι συνάδελφοι. Άδα βάσει του 123 του κανονισμού σας αποστήλαμε μια επεξήγηση για τη μελλοντική διαδικασία σε ό,τι αφορά τις γραπτές διακηρύξεις. Οι υπηρεσίες του Κοινοβουλίου συνέταξαν ένα περιεκτικότατο έγγραφο το οποίο και θα ε, διαβιβαστεί σε όλους τους συναδέλφους. Και τώρα να περάσουμε στην ημερήσια διάταξη. Στην ε, σημερινή στην τρονή φάση έχω μόνο μία αλλαγή να προτείνω. Για την ημερήσια διάταξη ζητάτε το λόγο. Κοιτάξτε, να ολοκληρώσουμε τα... τις ημερήσιες διάταξης και θα σα δώσω μετά το λόγο. Στην ημερήσια διάταξη